Doamnelor și domnilor, declar ședința Comisiei PETI deschisă. Doamnelor și domnilor, aș dori să doresc... Uh, Κυρίες και κύριοι, κηρύσω την έναρξη των εργασιών της συνεδρίασής μας, της συνεδρίασης της Επιτροπής Αναφορών και θέλω να Καλωσορίξω εξ ονόματός σας τον συνάδελφο Βαλέσα. Η κυρία Ματσόνη, πρόεδρος Επιτροπής μας, ε, δεν μπορεί να είναι εδώ την πρώτη ώρα της σημερινής συνεδρίασης, αλλά θα απουσιάζει και στη διάρκεια ενός μέρους της αυριανής συνεδρίασης γιατί υπάρχουν και συνεδριάσεις ταυτόχρονας Επιτροπής Ρέτζι. Υπάρχει μια αλλαγή στο σχέδιο ημερησιά διάταξης, συγκεκριμένα αφορά το σημείο 8. Κατόπιν αιτήματος ε, μελών της αντιπροσωπείας ε, θα αναβληθεί και το σημείο 5 θα το, συζητήσουμε αργότερα στην ε, ημερήσια διάταξη. Οι αναφέροντες και άλλοι προσκεκλημένοι θα είναι παρόντες για το σημείο 9. Life. Και για το σημείο 14, αναφορά 1327 του 2010, το σημείο 15, η αναφορά 161 του 2006, επίσης θα έχουμε παρουσία το αναφέροντο, συγκεκριμένα του κυρίου Ταν Μπρέναν και συναδέλφων αλλά και εκπροσώπων των Ιρλανδικών Αρχών. Για το σημείο 16, για την αναφορά 886 το 2005, θα έχουμε επίσης παρουσία για το 17, αναφορά 1518 του 2008, για το κυνήγι πτηνών, αγρίων πτηνών στη Βουλγαρία. Και σε ό,τι αφορά το σημείο 18 που αφορά το εμπόριο προϊόντων φώκιας θα έχουμε εκπροσώπους από το Human Society International. Θα ξεκινήσουμε την γνωμοδότηση για την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ύδατα. Έχουμε τον κύριο Χουντή, συντάκτη νομοδότησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κληθεί. Ο κύριος Μάρκο Κασπαρινέτη συγκεκριμένα είναι παρόν, εκπροσωπώντας την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά θα δώσω πρώτα απ' όλα το λόγο στον εισηγητή για να μας παρουσιάσει τη γνωμοδότησή του. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Επειδή είμαι καινούριο στην Επιτροπή, πείτε μου σας παρακαλώ πόσο χρόνο έχω για να μην κουράσω τους, τους παρόντες και παρούσες συναδέλφους. Πόσο χρόνο... Câte doriți, domnule raportor, as much as you like. Όσο χρόνο θέλετε. Here in the plenary, so you can talk as long... Δεν είμαστε στην Ολομέλη, άρα έχετε όσο χρόνο θέλετε. <laughs> <laughs> Το μικρόφωνο σας παρακαλούμε. επειδή οι ομιλίες μας στην Ολομέλεια είναι ενός λεπτού ή δύο λεπτών, θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται αναλυτικός αλλά και σύντομος για να μπορέσει να γίνει συζήτηση και να μην πέσει και έξω και το πρόγραμμά μας. Με χαρά ανέλαβα αυτή τη γνωμοδότηση. Σας θυμίζω ότι στην πρόσφατη Ολομέλεια, αγαπητοί συνάδελφοι, του Στρασβούργου ψηφίσαμε, εγκρίναμε το ψήφισμα για το Παγκόσμιο Φόρουμ. Εκεί υπογραμμίζω ότι εγκρίναμε ότι το νερό είναι κοινό πόρο τη ανθρωπότητας και ότι η πρόσβαση στο νερό είναι θεμελιώδες και οικουμενικό δικαίωμα. Εκεί εγκρίναμε ότι το νερό δεν πρέπει να αποτελεί πηγή κέρδους και για μένα και πιστεύω για όλους το νερό, ο αέρας είναι δημόσια αγαθά και είναι ανεκτήμητο αγαθό και πρέπει να το σεβόμαστε και να το διατηρούμε και η βιώσιμη διαχείρισή του αποτελεί αναγκαιότητα για το περιβάλλον και για την υγεία. Τα λέω αυτά γιατί αυτές οι βασικές μου πεπιθήσεις περιλαμβάνονται στο εισαγωγικό της γνωμοδότησης που ε, νομίζω ότι την έχετε διαβάσει. Επειδή το νερό είναι πανταχού παρόν, καθορίζει σε σημαντικό βαθμό το κλίμα και δεν μπορούμε να φανταστούμε τη ζωή χωρίς αυτό. Βεβαίως το θέμα ξεκινάει ότι ενώ είναι πανταχού παρόν δεν είναι πάντοτε εκεί που το έχουμε ανάγκη και στην κατάλληλη ποσότητα και στην κατάλληλη ποιότητα. Με αυτή την έννοια λοιπόν η οδηγία πλαίσιο για το νερό α, άπτεται των δύο αυτών πλευρών και τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα. Τέλος, σε σχέση με αυτά τα εισαγωγικά και με τη βοήθεια των ε, συνεργατών και με τη βοήθεια των εδώ υπηρεσιών Φαίνεται ότι από το 1988 υπάρχουν πολυάριθμες αναφορές στην Επιτροπή μας, στην Επιτροπή Αναφορών, σχετικά με το θέμα αυτό που αφορούν ε, σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οδηγία πλαίσιο λοιπόν για το νερό συνδυάζει τους στόχους τους ποσοτικούς, δηλαδή πόσο είναι διαθέσιμο, με τους στόχους τους οικολογικούς και τους ποιοτικούς, δηλαδή σε σχέση με την ποιότητα και ε, αντιμετωπίζει το θέμα της προστασίας των υδάτινων συστημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, καθορίζει μια σειρά από απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν μέσα σε καθορισμένες προθεσμίες, το υπογραμμίζω αυτό γιατί πρέπει να δούμε ποια είναι η πρόβλεψη, με στόχο να υπάρχει καλή οικολογική και χημική κατάσταση των υδάτων μέχρι το 2015. Στη γνωμοδότηση λοιπόν προσπάθησα να, να, να δείξω πέντε προβλήματα πέντε προβλήματα. Τα αναφέρω για την καλύτερη παρακολούθηση των όσων θα πω αναλυτικά για το καθένα μέσα στο πλαίσιο που σας υποσχέθηκα. Το πρώτο είναι η εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά από τα κράτη-μέλη. Το δεύτερο είναι η επάρκεια των υδάτινων πόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τρίτο είναι οι πηγές ρήπανσης. Το τέταρτο η σύγκρουση με άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές και η ανάγκη να ενσωματωθεί η πολιτική για το νερό σε αυτές και το πέμπτο, σημαντικό και αυτό, η συμμετοχή των πολιτών. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε την δέουσα, την πρέπουσα συμμετοχή των πολιτών σε μια πολιτική ευαισθητοποίησης και αντιμετώπιση του προβλήματος των νερών. Σε σχέση με το πρώτο, την εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο από τα κράτη, η εικόνα που έχουμε είναι ότι είναι άνηση τα κράτη μέλη την έχουν ενσωματώσει την οδηγία άλλα με καθυστέρηση άλλα εγκαίρως αλλά δείχνει ότι υπάρχει μια διαβάθμιση σε σχέση με τη διαχείριση και ότι η καλή οικολογική κατάσταση των υδάτων απέχει πολύ από τα αποδεκτά επίπεδα και τους στόχους. Σημειώνω εδώ ότι σε ένα πρόσφατο Euro workshop, που έγινε μια ημερίδα, μια ημερίδα εργασίας που οργάνωσε η Επιτροπή Περιβάλλοντος, η οποία έχει και την βασική ευθύνη για τη σύνταξη της έκθεσης, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ξεκάθαρα ότι οι κύριοι στόχοι της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά δεν ε, θα επιτευχθούν στις προθεσμίες που τίθενται. Εδώ προτίθεμε και από τη συζήτηση με τροπολογία να το κάνουμε πιο επίγον και να προτείνουμε τι πρέπει να γίνει ώστε να καλυφθούν ας το πούμε οι ημερομηνίε αφού η διαπίστωση, η πρώτη εκτίμηση είναι ότι δεν θα γίνει κατορθωτό. Το δεύτερο θέμα ε, έχει να κάνει με την επάρκεια των υδάτινων πόρων όπου σε ορισμένες περιπτώσεις στην Ευρώπη έχει φτάσει σε κρίσιμα επίπεδα. Και επειδή όταν μιλάμε για επάρκεια υδάτινων πόρων στην Ευρώπη καταρχήν το μυαλό μας πάει στη Νότια Ευρώπη θα σας έλεγα αγαπητοί συνάδελφοι ότι πρόβλημα υπάρχουν, υπάρχει και στη Βόρεια Ευρώπη ή να πούμε και σε περιοχές που οι βροχοπτώσεις είναι πιο άφθονες από τη Νότια Ευρώπη ή σε ορισμένες περιοχές. Ε, νομίζω ότι και στο Βέλγιο, στην Τσεχία, στην Πολωνία, τουλάχιστον με τα στοιχεία που διαθέτουμε, στη Βόρεια Ιταλία υπάρχουν προβλήματα. Βεβαίω υπάρχουν τα προβλήματα στι χώρε ή και περιοχέ που η λειψιδρία εμφανίζεται σε μόνιμη βάση και επηρεάζει συνολικά το πρόβλημα. Ισπανία, Νότια Ιταλία, Κύπρος και Μάλτα. Επομένως, επομένως, μια ορθολογική διαχείριση των υδάτων αφορά, που είναι αναγκαία αφορά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και επίγει η αναθεώρηση της πολιτικής σχετικά με το θέμα αυτό της λειψιδρίας και της ξηρασίας. Το τρίτο πρόβλημα από τα πέντε που προσπαθεί να αντιμετωπίσει η γνωμοδότηση είναι το θέμα της ρήπανσης, της ρήπανσης, τι ρηπαίνει το νερό. Ε, εδώ η καταγραφή λέει τα λίματα των αστικών περιοχών, η υγειονομική ταφή, τα βιομηχανικά και χημικά απόβλητα, τα φυτοφάρμακα αποτελούν ορισμένες από τις πιο συνήθεις αιστείες μόλυσης των υδάτων. Αυτό που ζητάμε, αυτό που ζητάω, αυτό που εισηγούμε να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να παράσχει μεγαλύτερη, περισσότερη υποστήριξη στην επεξεργασία των λιμάτων, εγκαταστάσεις κλπ και στις υποδομές των δικτύων αποχέτευσης στα κράτη-μέλη. Υπογραμμίζω επικουρικά στο σημείο αυτό ότι έχω ανησυχία, όπως φαίνεται και στην γνωμοδότηση, ότι στη νέα πρότασή της, η Κομισιόν, περιλαμβάνει μόνο 15 νέες χημικές ουσίες από έναν κατάλογο 2.000 δυνητικά επικίνδυνων ουσιών που πρέπει να παρακολουθούνται σε σχέση με τη σύνθεση και τη σύσταση του νερού και νομίζω ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος πρέπει αυτή την παράληψη να την υπογραμμίσει. Το τέταρτο και πρώτο τελευταίο σημείο είναι η σύγκρουση που έχουμε, αυξανόμενη σύγκρουση μεταξύ της πολιτικής των υδάτων με άλλες πολιτικές όπως η ενέργεια, η γεωργία, οι μεταφορές, η βιομηχανία, η αστική ανάπτυξη. Εκεί βλέπουμε εν της πράγμαση ένα θα έλεγε κανείς αρχέτυπο ένα βασικό δίλημα που εμφανίζεται πάντα αν η οικολογία είναι εναντίον της οικονομίας, οικολογία versus οικονομία. Δεν το εισηγούμεθα ότι έτσι είναι τα πράγματα γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει και μπορεί να βρεθεί ισορροπία μεταξύ και της προστασίας των οικονομικών των υδάτινων οικοσυστημάτων και των οικονομικών παραγόντων που πιέζουν προς την άλλη κατεύθυνση. Αναφέρουμε εδώ πιο αναλυτικά και έχει νομίζω την αξία το πρώτο, η ενέργεια, οι σημερινές κλασικές μορφές ενέργειας που χρησιμοποιούμε είναι οι πιο υδροβόρες, θα έλεγε κανείς, ε, πολιτικές, πολιτικές της ενέργειας. Ε, που καταναλώνουν σύμφωνα με τα στοιχεία η ενέργεια, οι κλασικές μορφές ενέργειας, το 45% των υδάτων που αντλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει εξ αυτής της διαπίστωσης η στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και μάλιστα αυτές που δεν σπαταλούν ή αξιοποιούν νερό είναι επίγουσα παραπάνω από άλλες φορές και εξ αυτού του λόγου και του θέματος που συζητάμε. Εδώ μπορούμε ε, να καταθέσουμε και πιο σχετική αυστηρία, ας το πούμε έτσι, τροπολογία. Και επίσης αναφέρομαι και στον τομέα της γεωργίας όπου υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν αναφορές για υπεράντληση των υδάτινων πόρων και για ρήπανση από τα φυτοφάρμακα. Εδώ υπάρχει το θέμα των επιδοτήσεων και των κριτηρίων. Ε, επιδοτήσεις σε υδροβόρες καλλιέργειες πρέπει να ξανακοιταχτούν παρά το γεγονός ότι υπάρχουν προβλήματα, δεν μπορείς από τη μια στιγμή στην άλλη να τα αντιμετωπίσεις. Θα μπορούσε εδώ να γίνει με μια πιο στοχοθετημένη, στοχοθετημένα κριτήρια και επίσης ε, η πρόθεσή μου είναι με μια τροπολογία να ζητήσουμε την ανακύκλωση του αστικού και του βιομηχανικού νερού και να διοχετεύεται σε καλλιέργειες και αναδασώσεις. Σε κάθε περίπτωση ε, θεωρώ ότι η ενσωμάτωση της πολιτικής για το νερό σε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές πρέπει να, να είναι καταγεγραμμένη. Και τελειώνω με το πέμπτο θέμα που σας υποσχέθηκα, που αναλύονται στη γνωμοδότηση και που είναι ότι πρέπει να εμπλακούν σε όλη αυτή τη διαδικασία οι Ευρωπαίοι πολίτες. Εδώ τι έχω να παρατηρήσω είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχει πλήρης πληροφόρηση των σχεδίων των, σε περιφερειακό, σε τοπικό επίπεδο, το τι σχεδιάζεται, το πόσο υδροβόρες είναι αυτές οι δραστηριότητες, με συνέπεια να μην μπορούν να παρέμβουν οι πολίτες, δεν υπάρχει πάντα η διαφάνεια. Επομένως και καταλήγω, νομίζω ότι πρέπει να ζητήσουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτιστούν επιγόντως, θα έλεγε κανείς, προγράμματα που να ευαισθητοποιούν τους πολίτες σχετικά με την εξοικονόμηση, μια κουλτούρα εξοικονόμηση και αποδοτική χρήση του νερού από το σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτά ε, θα ήθελα να σας ε, παρουσιάσω στα βασικά σημεία της γνωμοδότησης. Προφανώς ε, θα συνεργαστούμε, είμαι έτοιμο να συνεργαστώ και περιμένω και σχόλια, τροπολογίες για να καταλήξουμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ και πάλι κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χούντι, για την αναλυτική αυτή παρουσίαση. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριος Γκάσπαρη Νέτη, Μάρκο, εκπρόσωπος της Κομισιόν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει το σχέδιο γνωμοδότησης και την ποιότητα των συστάσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης. Σε ό,τι αφορά τα όσα είπε ο εισηγητής, ε, συμφωνούμε. Πέντε είναι τα βασικά θέματα και πράγματι πάνω απ' όλα ε, πρέπει να εφαρμοστεί η οδηγία πλαίσια για τα ύδατα. Γνωρίζετε ότι έω τα τέλη του τρέχοντο έτου θα αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Blueprint για τα ύδατα ε, τα περί τη εφαρμογή και στα τέλη του έτου αναμένεται η δεύτερη έκθεση για την εφαρμογή. Είναι δηλαδή μια χρυσή ευκαιρία αυτή για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διατυπώσει περαιτέρω σχόλια εφόσον το επιθυμεί. Σε ό,τι αφορά τα επιτεύγματα, δηλαδή το κατά πόσον έχουν επιτευχθεί περιβαλλοντικοί στόχοι και αν θα επιτευχθούν μέχρι το 2015, η κατάσταση ε, δεν είναι ομοιόμορφη στα κράτη-μέλη και αυτό εξηγείται από την θεμελιώδη διαφορά μεταξύ τη οδηγία για τα ύδατα αφενός και τη οδηγία για την ποιότητα του αέρα αφετέρου. Γνωρίζετε, φαντάζομαι, ορισμένοι από εσά ε, και τι δύο οδηγίε, ε, διότι και πολλέ αναφορέ σχετίζονται με αυτέ τι δύο οδηγίε. Διαφορετικά νομοθετήματα πάντω αφορά την ε, οδηγία για την ποιότητα του αέρα, παράταση ή παρέκκληση δίνεται μόνο εφόσον συμφωνήσει η Κομισιόν. Άρα υπάρχει και των προτέρων εξάντε έλεγχο ε, για τα αιτήματα παρέκκλησης ό,τι αφορά τις οριακέ τιμές για την ποιότητα του αέρα. Και όπως γνωρίζετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί με ιδιαίτερη αυστηρότητα όλα αυτά τα αιτήματα για παρεκκλήσεις, για εξαιρέσεις. Ό,τι αφορά τώρα την νομοθεσία για τα ύδατα, η κατάσταση είναι αντίστροφη θα έλεγα. Θα σας εξηγήσω με σωστή εννοώ. Τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να αναβάλουν την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων τις οδηγίες για τα ύδατα. Έχουμε μεν ε, την προθεσμία του 2015, αλλά στα ε, σχέδια διαχείρισης ε, λεκανών απορροής, τα οποία μελετούμε, βλέπουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις τα κρατη πιστεύουν ότι οι στόχοι δεν θα επιτευχθούν το 2015, αλλά το 2021 το νωρίτερο. Αυτό δεν είναι ικανοποιητικό. Είμαστε τώρα στη φάση της αξιολόγησης καθενός σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής. Τεράστιο βέβαια αυτό το εγχείρημα. Θα έχετε τα σχετικά στοιχεία στην έκθεσή μας και θα δείτε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Για το δεύτερο ζήτημα δεν έχω να προσθέσω κάτι σε σχέση με όσα προείπε ο εισηγητής. Τα θέματα το ποσοτικό δηλαδή. Ε, τώρα, στο θέμα της ε, ποιότητας και τη ρήπανση, ε, τους ρήπους ε, των υδάτων, πώς να σας το πω, βλέπω κάποια διαφορά στον τρόπο με τον οποίο ο εισηγητής ε, αντιλαμβάνεται την δραστηριότητα τη Κομισιόν και με τον τρόπο που εγώ την αντιλαμβάνω. Θα σα εξηγήσω τι εννοώ. Μιλήσατε, κύριε Σιγητά, για τι ουσίε προτεραιότητα. Μια οδηγία την οποία υπέβαλε πριν από κάποιε εβδομάδε η Κομισιόν, όπου έχει ορίσει ω προτεραιότητα 15 ουσίε. Ποιο είναι ο λόγο, Ο λόγο είναι ότι στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία εστιάζουμε σε αυτέ τι ουσίε προτεραιότητα, οι οποίε απαντούν στα περισσότερα ή σε όλα τα κράτη. Αλλά σε ό,τι αφορά την οδηγία πλαίσιο για τα είδωτα, Ξέρουμε ότι υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να συμπληρώσουν τον κατάλογο με οποιαδήποτε άλλη ουσία θεωρούν ότι είναι ε, σκόπιμο να συμπεριλάβουν για τη χώρα του. Άρα ο κατάλογο ουσιών προτεραιότητα που προτείνουμε εμεί σε καμία περίπτωση δεν είναι πλήρη, δεν είναι εξαντλητικό. Μπορεί δηλαδή να συμπληρωθεί από τα κράτη-μέλη αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο τοπικό πρόβλημα. Για το mainstreaming και την ολοκλήρωση Συμφωνώ απόλυτα, συμφωνεί και η Κομισιόν απόλυτα με τον εισηγητή για πιθανές συγκρούσεις, αντιπαραθέσεις με τη Γεωργία, παραδείγματο χάρη. Όλα αυτά πρέπει να επιληθούν και είναι θέματα τα οποία θα τα συζητήσουμε και στο πλαίσιο του blueprint. Για τη συμμετοχή τώρα των τον άρθρο 14, εκεί υπάρχει υποχρέωση των κρατών μελών για διαβούλευση. Έξι μήνες είναι η προθεσμία. Δράτω με τις ευκαιρίες για να αναφέρω ότι πριν από δύο ημέρες δρομολογήσαμε τη δημόσια διαβούλευση για το blueprint, όχι για το κείμενο βέβαια, αλλά τις γενικές επιλογές πολιτικής και οποιοδήποτε, οποιαδήποτε μη κυβερνητική οργάνωση κτλ. μπορεί να συμμετάσχει σε αυτή τη δημόσια διαβούλευση που ξεκίνησε πριν δύο ημέρε. Για το σχέδιο γνωμοδότηση τώρα, ε, δύο σχόλια έχω. Ελπίζω να μην καταχρώμε του χρόνου σα, θα προσπαθήσω πάρα πολύ σύντομο. Συμφωνούμε βέβαια με τα σημεία τα οποία αναφέρει ο εισηγητή και συγκεκριμένα με τις παραγράφους 4, 7 και 8 σε ό,τι αφορά την υποχρέωση των κρατών μελών να πετύχουν μια πολύ καλή περιβαλλοντική ε, κατάσταση. Αλλά μας ανησυχεί λίγο το ότι στο σχέδιο της γνωμοδότησης ε, το Κοινοβούλιο καλεί την ε, Κομισιόν ναι με να δείξει μεγαλύτερη αποφασιστικότητα σε ερευνές της, αυτό συμφωνούμε. Αλλά λέει μετά στο 9 συγκεκριμένο, ως εκ τούτου να έχει μια λιγότερο παθητική και συμβιβαστική στάση. Ε, δεν συμφωνώ με αυτή την ε, δήλωση. Δεν νομίζω ότι η Κομισιόν είναι παθητική και συμβιβαστική. Το κάθε άλλο στα θέματα των υδάτων. Αλλά για να τεκμηριώσω τη δήλωσή μου αυτή, θα σας δώσω κάποια στοιχεία για τις διαδικασίες επί οι οποίες ξεκίνησαν τα τελευταία δύο χρόνια. Γνωρίζετε ότι το περιβαλλοντικό δίκαιο είναι μια πολύ σημαντική πηγή ε, παραβάσεων εν γέννη και τα ύδατα στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας είναι και η μεγαλύτερη πηγή για παραβάσεις και για το 2010 και για το 2011. 713 υποθέσεις άνοιξαν το 10, 31% 31% επαναλαμβάνω φορούν τα νερά. Το 2011 908 υποθέσεις είχαμε και το 24% αυτών αφορούσε το νερό. Άρα θα ήθελα να αμφισβητήσω αυτή τη ε, διατύπωση του σημείου 9 ότι πρέπει να έχουμε μια λιγότερο παθητική και συμβιβαστική στάση. Ε, θα σας πω για τα κράτη-μέλη τι πιστεύουν για το αν είμαστε παθητικοί ή συμβαστικοί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση. Το κείμενο για πρώτη φορά τίθεται σε συζήτηση στην Επιτροπή μας. Παρακαλώ τους συναδέλφους να εκφράσουν τις παρατηρήσεις τους. Η κυρία Άουγκεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να μιλήσω δανέζικα σήμερα. Και πρώτα θέλω να ευχαριστήσω τον συντάκτη της γνωμοδότησης. Νομίζω ότι συμφωνούμε. Συμφωνώ στις εκτιμήσεις του. Καταλαβαίνω ότι η Κομισιόν ενοχλείται από την κριτική ότι τηρεί παθητική στάση. Αλλά και οι χώρες μέλη δεν κάνουν τίποτα. Ωραία είναι να δραστηριοποιείται η Κομισιόν, αλλά μετά δεν γίνεται τίποτα. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην κατανομή των κονδυλίων. Εμείς βλέπουμε εδώ να διαπιστώνουμε την αρχή του προβλήματος της λειψιδρίας που πάει να γίνει παγκόσμιο πρόβλημα. Θα αυξάνεται και η τεράστια ρήπανση των νερών και επίσης γίνεται μια τεράστια σπατάλη. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέπουμε για παράδειγμα στις τουαλέτες να χύνονται τέτοιες ποσότητες νερών και στην Δανία διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν τώρα τρόποι στα αυτόματα μηχανήματα που πλένουν αυτοκίνητα για κάθε πλήσιμο αυτοκινήτου να μην δαπανώνται πάνω από 4 λίτρα. Είναι δυνατόν. Χρειάζεται λοιπόν να γίνει πολύ μεγαλύτερη επένδυση σε πράσινες τεχνολογίες, τεχνολογίες εξοικονόμησης της ενέργειας αλλά και του νερού γιατί θα είναι εποφελής αμοιβαία και για τον άνθρωπο και για τη φύση η ε, κατάσταση αυτή οι καινοτομίες αυτές πρέπει να ενισχυθούν διότι δεν σημαίνει οι επενδύσεις αυτές μόνο επιβάρυνση των χωρών μελών αλλά μέσα σε αυτά κρύβεται και σημαντικές ευκαιρίες για την πρόοδο. Αυτά πρέπει να περιληφθούν στο κείμενό μας. Εγώ θα αρκεστώ σε αυτά για την ώρα και για τις χημικές ουσίες εγώ ήμουν εισηγήτρια στην προηγούμενη θητεία και είχαμε συζητήσει τότε για μια οδηγία για τα νερά της αποχέτευσης, των αποχετεύσεων. Εκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έδρασε με έπαρκη αυστηρότητα σε ό,τι αφορά δηλαδή την περιεκτικότητα σε διοκτώνα των διαφόρων αποβλήτων. Και στη Δανία και αλλού βλέπουμε ότι αυξάνεται σε τεράστιο βαθμό η χρήση των ζυζανιοπτών και λοιπόν. Και αυτά τα ζυζανιοκτώνα καταλήγουν στα υπόγεια νερά. Και τα υπόγεια νερά θα έπρεπε να τα προστατεύσουμε ως κόρυνο φθαλμού, διότι από εκεί αντλούνται τα πόσιμα ύδατα. Ας μην ασχοληθούμε με τον ορισμό του τι είναι υγιές νερό. Πρέπει να μιλάμε για καθαρό νερό. Και εκεί πρέπει να ισχύουν πάρα πολύ αυστηροί περιορισμοί, γιατί είναι πολύ σημαντικό ο τομέα αυτό. Ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κομισιόν κάνει πολλά πράγματα. Ξέρω όμω επίση ότι ε, ε, η Κομισιόν, έχει αντιληφθεί και αυτή ότι πολλέ χώρε δεν κάνουν τίποτα. Διότι συχνά και στη Δανία το ακούω αυτό. Αφού οι Γερμανοί κάνουν το Α, τότε και εμείς μπορούμε να κάνουμε το Α. Αν όμως οι εύπορες χώρες δεν λαμβάνουν επαρκή φροντίδα για το νερό, τι θα κάνουν άλλες χώρες λιγότερο εύπορες. Ε, συμφωνώ λοιπόν απόλυτα με τη γνωμοδότηση. Η Κομισιόν θα μπορούσε πράγματι να ασκήσει κάπως περισσότερη πίεση για την τήρηση των διατάξεων της οδηγίας. Ευχαριστώ. Vă mulțumim, doamna Ocan, pentru această prezentare. Dau în continuare cuvântul domnului Salavracos. ευχαριστούμε. Ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή για την έκθεσή του και εάν θα ήθελα να δηλώσω τις δικές μου προτεραιότητες για το μέλλον της Ευρώπης, ίσως και του πλανήτη, θα το έβλεπα ότι πρώτα έρχεται η καταπολέμηση της φτώχειας του κοινωνικού αποκλεισμού και του φαινομένου της ανεργίας, δεύτερο το περιβάλλον, μέσα στο περιβάλλον αντάσσεται και το θέμα νερό, και τρίτο δημογραφία και μετανάστευση. Αυτά είναι τα τρία, τρεις μεγάλοι τομείς και πολλοί άλλοι βέβαια στους οποίους πρέπει να επικεντρωθούμε και να μην παραμείνουμε ένα κλαμπ κοινωνικού προβληματισμού αλλά να προχωρήσουμε και σε δράσεις οι οποίες θα υλοποιήσουν τις σκέψεις μας και τον προβληματισμό μας πάνω στα θέματα αυτά. Ε, νομίζω ότι η έκθεση ε, αντιμετωπίζει με σωστό τρόπο το θέμα του ύδατος σαν κοινωνικού αγαθού και ε, από πλευρά μου θα έλεγα ότι θα ήθελα μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην εξασφάλιση των πηγών και των υπόγειων υδάτων τρόπον ώστε να μπορέσουμε να περισσώσουμε ό,τι είναι δυνατόν να περισσώσουμε σε συνδυασμό με το θέμα των ε, ε, αστικών λιμάτων τα οποία δυστυχώς έχουν αποδειχθεί ότι επιφέρουν τεράστια καταστροφή κυρίως στα υπόγεια ύδατα και δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα για την υγεία των ανθρώπων. Ε, σε γενικέ γραμμέ θεωρώ ότι είναι μια πολύ επιτυχημένη έκθεση και θα καλούσα και εγώ με τη σειρά μου την Κομισιόν, η οποία τη βλέπω έχει καλό προβληματισμό πράγματι, να δράσει με εντονότερο τρόπο διότι όλα αυτά θα τα δούμε μπροστά μας. Η λειψιδρία είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε τα προσεχή 5-10 χρόνια. Ε, πολλοί μιλάνε ότι ο επόμενος πόλεμος θα είναι ο πόλεμος του νερού σε ορισμένες περιοχές, ιδιαίτερα της Μέσης Ανατολής. Ε, να μην φτάσουμε ως εκεί. Πρέπει να κάνουμε δράσεις όμως. Το έχουμε εντοπίσει το πρόβλημα, να δράσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Mulțumim, Σας ευχαριστούμε. Εάν δεν υπάρχουν ε, άλλες παρεμβάσεις, παρακαλώ τον εισηγητή να ολοκληρώσει τη συζήτηση αυτή, εφόσον έχει να προσθέσει κάτι. Έχετε το λόγο, κύριε Χουντή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις και τον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Ε, τι θέλω να πω όπως φάνηκε από τη συζήτηση και οφείλω να σας πω ότι πίστηκα ακόμα περισσότερο σε, για ορισμένα σημεία που ισχυρίζομαι στη γνωμοδότηση και ίσως και με τροπολογίες να τα Το πρώτο ότι πρέπει, αφού οι προβλέψεις για την ενσωμάτωση και την εφαρμογή της οδηγίας ε, σε σχέση με τις προβλέψεις δεν είναι βίωνοι, πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να εφαρμοστεί. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη πίεση και στην Κομισιόν και στα κράτη-μέλη. Αν γίνεται κατανοητό η αξία, η σημασία που αναφέρθηκαν και άλλοι συνάδελφοι, θα πρέπει να υπάρξει ε, η μεγαλύτερη δυνατή πίεση. Ε, ε, εκεί θα έβαζα και τον τομέα πιο ενεργητική δράση, ούτως ώστε να υπάρξει εφαρμογή. Το δεύτερο που και κατά το ξεδίπλωμα της συζήτησης φαίνεται είναι ότι πρέπει να υπογραμμίσουμε το γεγονό ότι η πολιτική για το νερό πρέπει να σωματωθεί σε όλε τι ευρωπαϊκέ πολιτικέ. Ιδάλω δεν το αντιμετωπίζει. Θα το αντιμετωπίσει κάποια στιγμή όταν είναι θέμα της διάταξη και μετά θα το χάσει. Και αν το χάσει, δεν θα μπορέσει να το αντιμετωπίσει για μια σειρά λόγου που αναφέρθηκαν και που του γνωρίζουμε και στην πράξη σε σχέση με άλλε πολιτικέ που άπτονται τη ενέργεια κλπ. κλπ. Τώρα, ε, για ορισμένε παρατηρήσει. ε, που έκανε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν και τον ευχαριστώ για αυτό, θα ήθελα να πω ότι επιμένω στο σημείο πρώτο, στο σημείο για τις πηγές ρήπανσης. Θεωρώ ελλειπή την καταγραφή και την ε, αναζήτηση ή τον έλεγχο μόνο από 15 χημικές ουσίες με την έννοια ότι ίσως είναι ο κοινός παρονομαστής για όλες τις χώρες αν κατάλαβα καλά την τοποθέτησή του. Ε, θέλω να πω ότι όπως τονίστηκε και από άλλους συναδέλφους, ότι με την ανάπτυξη των φυτοφαρμάκων, της χημικής βιομηχανίας και των διάφορων άλλων σκευασμάτων και υλών που χρησιμοποιούμε καθημερινά, απορριπαντικά τούτο, με νέες ύλες, με νέες ουσίες, με νέες συνθέσεις στοιχείων, είναι φανερό ότι όλα αυτά, καθώς επηρεάζουν τα υπόγεια ύδατα κτλ. κάνουν πιο απαιτητικό, πρέπει να κάνουν πιο απαιτητικό τον έλεγχο και επομένως ε, νομίζω ότι πρέπει να συμπληρωθεί αυτός ο κατάλογος και να μην μένει μόνο στα 15 στοιχεία. Εν δυνάμει είναι 2.000, δεν ξέρω αν μπορεί να τα περιλάβει όλα. Αν τα αφήσουμε σε επίπεδο εθνικής νομοθεσίας, εκεί το φοβάμαι το θέμα. Δεν ξέρω για ποιους λόγους μπορεί να μην ε, είμαστε απαιτητικοί ως προς αυτό. Υπάρχει και μια δυναμική στην, στις πηγές αυτό θέλω να πω, της, ε, ε, του νερού. Και για το τελευταίο, ε, εξαιρετικά κατατοπιστικό ήταν ε, σχετικά με το αν ε, η, περιβαλλοντική νομοθεσία παραβιάζεται και έχουμε μια μείωση σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έδωσε ο πρόσωπος της Κομισιόν για τις παραβιάσεις σε σχέση με τα νερά από 31 σε, από τα νερά στο 24. Αυτό αν δεν το δούμε συγκριτικά δεν σημαίνει κατά ανάγκη πως έχει βελτιωθεί η πολιτική για τα νερά. Μπορεί να έχει αυξηθεί, η δική μου εικόνα είναι αυτή, ότι έχει αυξηθεί στη διαχείριση των απορριμμάτων η παραβίαση το είχαμε συζητήσει πολλές φορές. Επομένως μπορεί συγκριτικά με τα νερά να έχει, βελτιωθεί, να έχει αυξηθεί των απορριμμάτων και τα νερά να έχουν μειωθεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως έχει βελτιωθεί γενικώ η κατάσταση ή ότι δεν έχουμε παραβιάσεις. Άλλωστε η αφορμή αυτής ή και η δική μας γνωμοδότηση ξεκινάει από το ότι έχουν έρθει χιλιάδες αναφορές από το 1988 όσο αφορά το σχετικό θέμα. Α, και επομένως και με αυτό το στοιχείο ε, επιμένω στην τοποθέτηση για την παθητικότητα της Επιτροπής σας ενισχυθεί η δραστηριότητά της παραπάνω και θα βρούμε τη διατύπωση την τελική αλλά επιμένω ότι η δική μας τοποθέτηση πρέπει να έχει έτσι ένα κριτικό σημείο και ένα απαιτητικό από την Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να υπενθυμίσω την προθεσμία για την κατάσταση τροπολογιών 28 Μαρτίου λίγη η προθεσμία. Και περνούμε στη συζήτηση των αναφορών που έχουμε στην Μεσιά Διάταξη. Η αναφορά 195 το 2011 θα συζητηθεί λίγο πιο μετά. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 6, την αναφορά 93 του 2011. Έχει κατατεθεί από τον Κλοντ Κόστ, εξ ονόματος της Ένωσης κατά των πλημμυρών, την ε, προστασία των υδάτων και, του περιβάλλοντος, και το περιβάλλον. Αφορά την επεξεργασία των νεκρών όμβριων υδάτων για την προστασία των επιφανειακών υδάτων στη Γαλλία. Δεν είναι παρόν αναφέρον. αλλά μπορούμε να ακούσουμε στα ακουστικά μας την ομιλία του. Θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτα απ' όλα, γιατί δεν έχουμε ακόμα στη θέση μας την ομιλία του αναφέροντος. Πρόσωπος λοιπόν της Κομισιόν έχει το λόγο. Το πρόβλημα που προκύπτει από την μη επεξεργασία των νερών της ροχής που πέφτουν των, όμβριων, των νεκρών των όμβριων υδάτων δηλαδή δεν έχει ληφθεί υπόψη επαρκώς. Για τα κράτη-μέλη υπάρχει υποχρέωση να λαμβάνουν μέτρα ώστε οι παραθαλάσσιες περιοχές να μην επηρεάζονται από την εκροή όμβριων υδάτων που δεν έχουν τύχη επεξεργασίας. Υπάρχει και ειδική οδηγία που περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις για την επεξεργασία που πρέπει να επιφυλάσσεται στα όμβρια ύδατα που φτάνουν με απρόσμενο τρόπο και που δεν καθίσταται δυνατό καθίσταται δυνατό να τύχουν ε, επεξεργασίας. Υπάρχει η, στα αγγλικά Float Directive που επιβάλλει στις χώρες μέλη να λαμβάνουν μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι οι κίνδυνοι από αυτά τα όμβρια ύδατα θα μειώνονται σε επίπεδο που να μην επηρεάζεται σημαντικά το περιβάλλον. Θα ήθελα ωστόσο να επιστήσω να επιστήσω την προσοχή σας σε δύο είδη εγκαταστάσεων που ενδεχομένως να υποστούν προβλήματα, να, να αντιμετωπίσουν προβλήματα είναι οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερών και επίσης και αποβλήτων. Στις σχετικές οδηγίες της Ένωσης που απαιτούν από τις χώρες μέλη να λαμβάνουν μέτρα είτε για την επεξεργασία των νερών είτε για την επεξεργασία των απορριμμάτων είναι σαφές ότι υπάρχουν, περιλαμβάνονται υποχρεώσεις που να διασφαλίζουν ώστε εάν ποτέ φτάσουν σε μεγάλες ποσότητες όμβρια ύδατα στις εγκαταστάσεις αυτές να μην επηρεαστεί η λειτουργία των εγκαταστάσεων. Λέγεται λοιπόν καθαρά, διατυπώνεται καθαρά ότι οι εγκαταστάσεις αυτές είτε των αστικών λιμάτων δηλαδή είτε των απορριμμάτων πρέπει να είναι κατασκευασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα, οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από την έλευση μεγάλων ποσοτήτων όμβριων υδάτων που δεν θα έχουν γίνει αντικείμενο επεξεργασία. Η Κομισιόν επιθυμεί να είναι σύντομη. Αντί να ζητήσει την λήψη νέων νομοθετικών μέτρων, η Κομισιόν θεωρεί ότι είναι προτιμότερο για την ώρα να εφαρμοστεί καλύτερα ισχύουσα νομοθεσία. Αυτά λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, από πλευράς της Κομισιόν. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Βασέσκο. Νομίζω ότι έχουν οι διερμηνείς στο κείμενο της ομιλίας του αναφερομένου. Α, το έχουν μόνο στα γαλλικά και παρακαλείται η γαλλική καμπίνα να αναγνώσει το κείμενο. Είναι πρωτότυπη η διαδικασία αυτή, λέει η κυρία Πασέσκου, αλλά σας παρακαλώ να προσπαθήσετε. αναφορά κάποιος διακόπτη δεν ακούτε ωραία λοιπόν αναφορά κατά της απόρριψης τον Ιανουάριο 2011 από το, από το Υπουργείο συγγνώμη, Περιβάλλοντος για την υποχρέωση επεξεργασίας των όμβριων υδάτων. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι μέλη της Επιτροπής Αναφορών, η επιστολή που απέστειλα στις 22 Ιανουαρίου 2011 περιλαμβάνει γεγονότα αδιαμφισβήτητα και ε, σχετικά με την όλο και αυξανόμενη ρήπανση της Μεσογείου για διαφόρους λόγους, αλλά για 99% προέρχεται από ύδατα που καταλήγουν στην ε, θάλασσα από τους ποταμούς. Βρισκόμαστε στην κατάσταση αυτή η οποία ε, επιδεινώνεται κάθε χρόνο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να παραμείνει αδρανές εν προκειμένου και να αναμένει απλώς μια βελτίωση. Είναι απαραίτητο να ληφθούν αποφάσεις με άμεσο αποτέλεσμα οδηγίες ή άλλα κείμενα. Με την ελπίδα ότι η έκκλησή μας αυτή θα γίνει, θα ε, γίνει δεκτή από πλευρά σας, σας παρακαλώ να δεχτείτε τα ειλικρινή μου στήματα. Ε, Ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Μπασέσκου. ο εισηγητής θα πρέπει να περιλάβει στο κείμενό του το κείμενο των αναφερομένων. Δεν υπάρχει αίτηση λήψεως του λόγου από την αίθουσα. Η κυρία Άουκεν ζητεί, σηκώνει το χέρι. Έχετε το, το λόγο, κυρία Άουκεν. Θέλω να μου πείτε να πω λίγα λόγια. Ε, κυρίως στις πόλεις, ε, το τι θα κάνουμε ε, στο μέλλον με τα όμπρια ύδατα. Νομίζω λοιπόν ότι σε πάρα πολλές ε, περιοχές, τον Ιούλιο ας πούμε στην Κοπενχάγη, δεν είχαμε καθόλου βροχές. Δεν αρκεί μόνο να κατασκευάσουμε ένα σύστημα που να διώχνει τα όμβρια είδωτα, πιο ε, λογικό θα ήταν να δημιουργήσουμε κάποιες δεξαμενές ε, στη στέγη ή κάπου αλλού, να μαζεύει τα όμβρια είδωτα, τα νερά της βροχής. Να συνεργαστούμε με αυτούς ε, που δημιουργούν τις αποχετεύσεις, τους υπονόμους, για να διαφυλάσσονται, να συγκεντρώνονται τα είδατα, Να προσπαθούμε να προσπαθήσουμε να δούμε πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Γίνονται λοιπόν πάρα πολλές ε, δουλειές πάνω σε αυτό, πολλές ε, σκέψεις και μελέτες και ξέρετε έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες εάν ε, εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτή την προετοιμασία, δηλαδή να προσπαθήσουμε να αποθηκεύσουμε το νερό αντί να το εκβάλουμε, να το αποδιώχνουμε γιατί είναι δαπανηρή όλη αυτή η διαδικασία. Αν λοιπόν ακολουθήσουμε αντίστροφη και διαφορετική διαδικασία, αυτό είναι πιο σωστό. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να καταρτήσουμε μια στρατηγική για να εξοικονομήσουμε νερό και να σώσουμε και τις πόλεις, να μην τις αφήσουμε να υποφέρουν από τη λειψιδρία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Άουκεν, αλλά βλέπω ότι και ο κύριος Γιάρα επιθυμεί να λάβει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κοιτάξτε, νομίζω ότι είμαστε μπροστά σε ένα δίλημα. Αν κατάλαβα καλά την απάντηση της Επιτροπής, χρειαζόμαστε... Δεν χρειάζεται να ανταποκριθούμε στο αίτημα του ετούντος, διότι αρκούν, αρκεί η κείμενη νομοθεσία, η ευρωπαϊκή. Ε, αναφέρεται ότι η προστασία των υδάτων ε, μέσα από την οδηγία πλαίσιο περί υδάτων ε, και την στρατηγική που ακολουθείται ρυθμίζεται αυτή η ανάγκη. Δηλαδή, από νομική σκοπιά δεν χρειάζεται να ικανοποιήσουμε το αίτημα του ετούντος γιατί ήδη ικανοποιείται. Το πρόβλημα όμως που υπάρχει και εδώ πραγματικά θεωρώ ότι η Κομισιόν έχει δίκιο, δηλαδή δεν θα βελτιωθεί η κατάσταση στην πρακτική με το να θεσπίσουμε άλλη μία νομοθετική πράξη. Και νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε την εξή πρόταση. Να πούμε στον Ετούντα ότι όσον αφορά το συγκεκριμένο αυτό αίτημά του να επιβάλλεται η απομάκρυνση υδάτων δεν χρειάζεται να ικανοποιηθεί αυτό το αίτημα γιατί είναι ικανοποιητική η κείμενη ισχύουσα νομοθεσία και μπορούμε βέβαια να παρακαλέσουμε και τον ετούντα να μας αναφέρει συγκεκριμένα παραδείγματα όπου κατά την δική του άποψη δεν ε, εφαρμόζεται η νομοθεσία. Ίσως ε, αυτός να είναι ο σωστός δρόμος. Εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Η Κομισιόν λέει αρκεί η κείμενη νομοθεσία και ο ετών επιθυμεί να θεσπιστεί να θεσπιστούν περαιτέρω νομοθετικέ ε, πράξεις. Αυτό όμω δεν θα βοηθήσει τίποτα στην πρακτική εφαρμογή. Εγώ ε, εντάξει, αν θέλετε να αφήσουμε ανοιχτή την ε, έτσι, ας την αφήσουμε, δεν με ενοχλεί. Αλλά κανονικά πρέπει να την κλείσουμε. Γιατί αν έχει συγκεκριμένε ενδείξει για συγκεκριμένε περιοχέ ότι τα πράγματα δεν λειτουργούν και δεν πάνε καλά, α μα το ε, πει και θα δούμε. Ευχαριστώ. Wortmeldung Κύριε Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μια κουβέντα θα ήθελα να πω σε σχέση με κάποιες νήξεις που έκανε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Υπάρχει σε αρκετές περιπτώσεις η περίπτωση που έχουμε όμβρια ύδατα που περνάνε μέσα από εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων με συνέπεια έχω πάρα πολλά παραδείγματα τουλάχιστον από την ελλάδα είναι από τα πιο μεγάλα προβλήματα με συνέπεια να ρηπαίνονται ευρύτατε θαλάσσιες περιοχές διότι περνάνε από τέτοιες εγκαταστάσεις. Επομένως, πάρα πολλά παραδείγματα. Επομένως, ενώ υπάρχει σχετική κοινοτική νομοθεσία, κατά την εφαρμογή ή και την, ε, την ε, δημιουργία τέτοιων εγκαταστάσεων κλείνουν τα μάτια, οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι ελλειπείς με πρόδειλα σφάλματα και η κατάσταση πάει να αντιμετωπιστεί εκ των υστέρων, αλλά η ζημιά έχει γίνει. Επομένως δεν φτάνει η, επίκληση νομοθεσίας, τουλάχιστον στην προκειμένη περίπτωση, ε, απαιτείται και η αυστηρή εφαρμογή. Άρα υπάρχει θέμα, δεν ξέρω αν θα πρέπει να μείνει ανοιχτή, υπάρχει τέτοιο θέμα και από αυτή την πλευρά ότι έχουμε να προστατευτούν οι θαλάσσιες περιοχές παραλίες της Μεσογείου, τουλάχιστον αυτό λέει η δική μου εμπειρία. Αυτό ήθελα να προσθέσω σε σχέση με την αναφορά που ακούσαμε κατά τον πρωτότυπο τρόπο. Κατά τα άλλα που θα μπορούσε να ήταν πιο ζωντανό αν ήταν εδώ και ρωτούσαμε κάτι πιο συγκεκριμένο. Um... În lumina comentariilor făcute, uh, consider totuși că această petiție... ευχαριστούμε πολύ. Παρακολουθήσαμε, <laughs> τις, ακούσαμε τις παρεμβάσεις αυτές προσεκτικά. Θεωρώ ότι πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Ας περάσουμε στο υπαριθμό, ή μάλλον ας επανέλθουμε στο 5, αναφορά 195 του 11, Εσείς κύριε Γιάρ. Να είμαστε διακόπτη. Ε, ναι, έχω το μικρόφωνο, ναι, ναι, ανοιχτό είναι. Αναμένω είναι. Να είμαστε έντιμοι και να αποστείλουμε ε, μια επιστολή στον αναφερόμενο, να μην χαθεί η αναφορά, αλλά να τη συμπληρώσει με συγκεκριμένα στοιχεία. Σημειώνουμε την παρατήρησή σας και προχωρούμε στην 195 και το λόγο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κ. Ερνάντες Λούκε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, το πρώτο που θέλω να υπογραμμίσω είναι το εξής. Με βάση τη διαχειριστική αρχή του προγράμματος με χώρα της από το 2000 2006 υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα όπου πήραμε 2.300.000 ευρώ και αυτό αυτό το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε ε, με ευρωπαϊκή συμμετοχή. Το σύνολο της δαπάνης και της επένδυσης ήταν ύψους 5 εκατομμυρίων χιλιάδων Λοιπόν, το σύνολο της επένδυσης ανήλθε σε 5.971.013 ευρώ. Από το 2007 και εντεύθεν το πρόγραμμα δεν χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 235 κάθετος 2004 και 186 κάθε 2006 της 28 Ιουνίου και της 18 Δεκεμβρίου του 2007 αντίστοιχα. Τα προγράμματα της ε, γεωργικής ανάπτυξης εγκρίνονται από την Επιτροπή αλλά ε, εκτελούνται από τα κράτη-μέλη. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι η χρηματοδότηση αυτού του προγράμματος που στηρίξαμε, τούτο εμπίπτει στις αρμοδιότητες της διαχειριστικής αρχής του προγράμματος και αυτό συμβοδίζει με την αρχή της ε, επιμερισμένης ε, διαχείρισης άλλες πληροφορίες για αυτό το Σεγκάν Αλγαρίγες, ε, ε, το πρόγραμμα της υδροδότησης, ε, θα πρέπει άλλες πληροφορίες, αν θυμείτε, να τις ζητήσετε από τις εθνικές αρχές. Και θέλω να υπογραμμίσω ότι το έργο αυτό είναι ανεξάρτητο από ένα άλλο πρόγραμμα για το οποίο οι Ισπανικές αρχές υπέβαλαν αίτημα χρηματοδότησης στο Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο. Και τα δύο αυτά έργα είναι ανεξάρτητα ε, και δεν συνδέονται μεταξύ τους. Ούτε σε επίπεδο σύλληψης, ούτε με οποιαδήποτε άλλη μορφή. Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Ράνθ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Να καλωσορίσω τους συναδέλφους μας ε, στην Επιτροπή Αναφορών. Ε, ορισμένους σα γνωρίζω από την Επιτροπή Γεωργίας. Έχω έρθει σε επαφή και από την Επιτροπή Γεωργίας με τους αναφέροντες και από το Γεωργικό Ινστιτούτο Σαν Ισίδρο της Καταλωνίας. Ε, τους είχα ζητήσει να έρθουν στην Επιτροπή μας. Συμφωνούμε με τα όσα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πράγματι δεν υπάρχει πρόβλημα χρηματοδότησης των δύο αυτών έργων. Σε αυτό συμφωνούμε. Όμως, η πρωτοβουλία αυτή πρέπει να παραμείνει, παραμείνει ανοιχτή, διότι δεν συμφωνούμε με αυτό που είπε η Κομισιόν ή που έχουν πει οι Ισπανικέ Αρχέ ότι είναι ανεξάρτητα τα δύο έργα αυτά. Όχι, δεν είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Θα σα πω γιατί. Ένα φράγμα μόνο υπάρχει για την έγκριση. Ε, λέγεται ότι είναι ένα φράγμα για άρδευση. Και έπειτα βασίζεται σε κονδύλια αποκλειστικά διατηθέμενα σε γεωργικέ δραστηριότητε. Κάποια δεδομένη χρονική στιγμή, οι Ισπανικές Αρχές συγκεκριμένα της ε, αυτόνομης περιφέρειας ε, της Καταλωνίας αποφάσισαν ότι αυτό το κανάλι ε, θα χρησιμοποιείται όχι μόνο για άρδευση αλλά και για δροδότηση. Και εκεί υπάρχει το πρόβλημα γιατί χάνεται η αρχική ιδέα. Δεν είναι ότι ένα μικρό μέρος θα πηγαίνει για την υδροδότηση, αλλά, για την αλλά ουσιαστικά δεν εξυπηρετεί πλέον τη γεωργία αυτό το κανάλι και έχει να κάνει με ε, έργα υδροληψίας και υδροδότησα. Πρέπει όμως ε, να τα έχουμε όλα υπόψη μας και τη γεωργία και την υδροδότηση των πόλεων. Δεν μπορούμε όμως να παραβιάζουμε ε, τα δικαιώματα των γεωργών της περιοχής αυτής της Σεγαργαρίγες. Δεν μπορούμε να στερούμε υπηρεσίες που είναι πάρα πολύ απαραίτητες για τις πόλεις. Γι' αυτό και το Γεωργικό Ινστιτούτο Σαν Ισίδρο της Βαρκελόνης θέλει να έρθει εδώ και να εξηγήσει ότι αυτά τα οποία λένε οι Ισπανικές αρχές, οι αρχές παραλαμβάνω της Περιφέρειας Καταλωνίας δεν ανταποκρίνονται, δεν αντιστοιχούν με τις αρχές του σχεδιασμού, της μελέτης για τη δημιουργία αυτού του καναλιού. Και γι' αυτό ναι, μεν αυτοί θεωρούν την Επιτροπή Αναφόρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να του ακούσει, του αναφέροντε δηλαδή, να καταλάβει του λόγου για του οποίου υποστηρίζουν ότι δεν είναι ανεξάρτητα μεταξύ του τα δύο έργα όπω ε, υποστηρίζουν οι Ισπανικέ Αρχέ. Ναι, δεν είναι θέμα χρηματοδότηση, είναι όμω θέμα θεμελιωδών δικαιωμάτων των ανθρώπων αυτών που θεωρούν ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά του από του υπεύθυνου τη αυτόνομη περιφέρεια τη Καταλωνία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Ράνθ. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θέλουν το λόγο. Η κυρία Άουκεν. Είναι δύσκολο να το παρακολουθήσει κανείς αυτό. Από ό,τι καταλαβαίνω, το πρόβλημα είναι πρόβλημα νομιμότητας. Δηλαδή, να περιλαμβάνεται αυτό το έργο σε ένα πρόγραμμα ε, χώρου τοποθεσίας Natura 2000. Αυτό, αυτό είναι που αμφισβητεί ο αναφερόμενος. Μα είναι μες στο κείμενο, κύριε Ράνθ. Την αναφορά διαβάζω. Γιατί τελώ εν συγχύσει. Εφόσον συγκρίνω το τι περιλαμβάνεται στην αναφορά και το, αυτά που άκουσα από την απάντηση, δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Αν μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει γιατί λαμβάνω μια τελείως διαφορετική απάντηση από αυτή που διάβασα στην αναφορά. Κοιτάξτε, και εγώ το ίδιο ερώτημα έχω όπως η συνάδελφός μου. Ίσως μπορεί κάποιος ε, να μας εξηγήσει έτσι με απόλυτη ηρεμία και ξεκάθαρα ε, περί ακριβώς πρόκειται όσον αφορά ε, αυτή την αναφορά τα μπερδέψαμε κάπως. Ε, ίσως λοιπόν κάποιος μπορεί ε, ήρεμα, αργά και καθαρά να μας εξηγήσει περί τίνος πρόκειται. Κυρία Εράνθε, ευχαριστώ. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Και εγώ ε, δεν το είχα καταλάβει πολύ καλά. Θέλω να σα πω το εξή. Σε καμία περίπτωση το Σαν Ισίδρο, το Γεωργικό Ινστιτούτο αυτό τη Καταλωνία, δεν θέτει υπό αμφισβήτηση ότι πρέπει να εφαρμόζονται τα αυστηρότερα δυνατά περιβαλλοντικά πρότυπα για ζώνε ειδική προστασία, πτηνών κτλ. Το αντίθετο χαίρονται πάρα πολύ και αυτό επιδιώκουν, να τηρεί την νομιμότητα. Και δεν υπάρχει και άλλος ε, τρόπος από την που ζητεί τη δημόσια χρηματοδότηση. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα που βλέπουμε εδώ έχει να κάνει με τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων εκείνων που επένδυσαν χρόνο, προσπάθεια, χρήμα για να επιτύχουν την άρδευση αυτή για την περιοχή σε γάρα Και από τη στιγμή που κατασκευάστηκε αυτή η δεξαμενή, αυτό το κανάλι, πώς να το πω, για να συγκεντρώνονται εκεί τα ύδατα εκείνα τα οποία προορίζονταν για τη γεωργία. Η δημόσια διοίκηση της αυτόνομης ε, περιφέρειας της Καταλωνίας αποφάσισε να τους στερήσει αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα που έχουν και να επαναχρησιμοποιήσει τα ύδατα αυτά στο μεγαλύτερο μέρος τους για την υδροδότηση και όχι για την άρδευση των ε, αγροτεμαχίων των ε, αγροτών αυτών που είναι στο Γεωργικό Ινστιτούτο αυτό σαν δεν θέτουν υποαμφισβήτηση τα περιβαλλοντικά πρότυπα. Το αντίθετο παραλαμβάνω, τα σέβονται, τα τηρούν και το έχουν αποδείξει. Όπω κάνουν και με όλα τα περιβαλλοντικά πρότυπα για την ε, προστασία φυσικών πάρκων, ε, χώρων που ε, περνούν πτηνά κτλ. Αλλά εδώ μιλάμε για κάτι άλλο. Αποφασίζει η Ισπανική Δημόσια Διοίκηση να του αφαιρέσει ένα δικαίωμα που είχαν και να αλλάξει τη χρήση αυτού του καναλιού που δεν προορίζεται πλέον για την άρδευση, αλλά υδροληψία και υδροδότηση πλέον. Και το λέω γιατί δεν είναι ξεκάθαρο καθόλου το θέμα και γίνεται μια προσπάθεια σύγχυσης να ανακατευθούν κάπως τα θέματα μεταξύ τους και γι' αυτό λέω να παραμείνει ανοιχτή αναφορά. Να ακούσουμε τους αναφέροντες, γιατί θέλουν να ε, μπορούν να απολαύουν το δικαιώματό του να μπορούν να ασκούν τη μεγιορική τους δραστηριότητα, που έχουμε ε, σε αυτή την περίοδο τόση κρίση, τόση οικονομικά προβλήματα. Λοιπόν, δεν μπορούν να του στερούν αυτό το δικαίωμα. Ε, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σα, κύριε Άικεν. Κοιτάξτε, δεν αρκεί η αιτιολόγηση αυτή. Δεν είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Η γεωργία τραβάει πολύ νερό. Και τότε βέβαια υπάρχει σπάνιδα νερού. Αυτό θα γίνει ξανά και ξανά. Και να πείτε ότι ε, πάντα το κάναμε αυτό, μπορούμε να πάρουμε το νερό από αλλού, μα τότε σύντομα θα καταλήξετε σε πόλεμο. Εγώ από αυτά που διαβάζω εδώ, δείχνουν ότι δεν δέχονται ότι χρειάζεται κάποιος περιορισμός στη χρήση του νερού. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Χρειάζεται μια καλύτερη παρουσίαση του θέματος. Από ό,τι διαβάζω εγώ την αναφορά και ακούω και κυριάζω και την απάντηση μάλιστα, όχι αυτή που άκουσα πριν, δεν θεωρώ ότι πρόκειται για αναφορά που μπορούμε να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε. Ίσως βέβαια έχω παρανοήσει όλη αυτή την ιστορία, αλλά είμαι υποχρεωμένη να δω αυτά που έχω μπροστά μου και που διαβάζω. η Προεδρεύουσα. Ακούσαμε τα επιχειρήματα και πρέπει να εξετάσουμε την αναφορά. Νομίζω ότι το καλύτερο είναι η αναφορά να παραμείνει ανοιχτή. Και το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη λοιπόν είναι η ογνωμοδότηση με θέμα 20 βασικότερες ανησυχίες των πολιτών της ενιαίας αγοράς. Το υπαριθμό 7 δηλαδή. ο κ. Γιάρ. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε του αναφερόμενου, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε. Έχει γίνει αίτηση για ένα έργο, τώρα για δύο, που τραβάνε νερό από την ίδια πηγή. Δεν μπορεί να γίνει διάλογος παρά μόνο με παρουσία των αναφερομένων. Και εάν κατάλαβα καλά, εάν πρόκειται για δύο έργα τα οποία πρόκειται να γίνουν θα χρειαστούμε εκπροσώπους και των δύο έργων. Οι δεμοί θα βρισκόμαστε διαρκώς σε σύγχυση. Φαίνεται να υπάρχουν σημαντικές συγκρούσεις συμφερόντων που δεν μπορούμε τώρα να κρίνουμε και να τάμουμε με τα λίγα έγγραφα που έχουμε στη διάθεσή μας. Να έλθουν λοιπόν εδώ την επόμενη φορά. Και αν κατάλαβα καλά πρόκειται για δύο έργα και αν κατάλαβα καλά ότι πρόκειται για δύο έργα το ένα είναι η χρήση των υδάτων για τη γεωργία, το άλλο είναι για ε, πόσιμο νερό, χρειαζόμαστε λοιπόν εκπροσώπου και των δύο πλευρών. Γιατί αλλιώ δεν πρόκειται να μπορέσουμε να βγάλουμε άκρη. Σα ευχαριστώ πολύ. Έχετε δίκιο κύριε Γιά. Και αυτό είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους επιθυμώ να διατηρηθεί ανοιχτή η αναφορά αυτή. Έρχομαι τώρα πάλι στο 7 με θέμα 20 βασικότερες ενισχύσεις των πολιτών και επιχειρήσεων για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Αρμόδια είναι η Επιτροπή Προστασίας των Καταναλωτών και συντάξει των Ομοδοτήσεων είναι ο κ. Μπουσούτιλ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή η γνωμοδότηση ε, προετοιμάστηκε για την ε, Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και αφορά την έκθεση που δημοσίευσε η Επιτροπή τον Αύγουστο του προηγούμενου έτους. Ε, πρόκειται λοιπόν για μία άποψη των πολιτών και των επιχειρήσεων και περιλαμβάνει η γνωμοδότηση αυτή, η έκθεση αυτή, 20 βασικές ανησυχίες. Η δική μας Επιτροπή καλύτερα να γνωμοδοτήσει και υπάρχει δυστυχώ χρονικό περιορισμό. Είναι και μακροσκελή η έκθεση. Γι' αυτό εγώ θα εστιάσω την προσοχή μου στα θέματα εκείνα τα οποία ε, πραγματικά έχουν σημασία για την Επιτροπή μα. Στη δική μου λοιπόν τη γνωμοδότηση καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριλάβει στις μελλοντικές της εκθέσεις ε, τα αποτελέσματα αναφορών που κατατίθενται στην Επιτροπή μας ε, και να ε, δώσει ιδιαίτερη σημασία στο δικαίωμα των πολιτών να αναφέρονται μέσω της Επιτροπής μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, ε, επισημαίνω τη σημασία του να γίνεται καλύτερη χρήση της διαδικασίας έτσι ώστε να βελτιωθεί η ε, νομοθετική διαδικασία και να ε, βελτιωθεί η συνειδητοποίηση για το δικαίωμα αναφοράς, κατάθεση αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο δεν είναι ένα δικαίωμα το οποίο δίδεται στους πολίτες μέσω της ε, Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κάτι άλλο που αναφέρω στην έκθεσή μου είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει στο μέλλον να συμπεριλάβει αναφορές στους βασικούς νόμους που έχουν σε σχέση με τις ανησυχίες των πολιτών. Και με τον τρόπο αυτό θα ε, δώσει θα διασαφηνεί την κατάσταση ε, σε σχέση με τις ανησυχίες των πολιτών και των επιχειρηματιών. Και με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθεί η συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πολίτες θα συνειδητοποιήσουν καλύτερα ε, τον τρόπο με τον οποίο σχετίζονται τα προβλήματα και οι λύσεις με συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και τέλος, κυρία Πρόεδρε, προσπάθησα στη γνωμοδότησή μου ε, να δώσω έμφαση να προβάλλω μεμονωμένες υπηρεσίες που προσφέρονται στους πολίτες. Πολλές ε, υπηρεσίες είναι χρήσιμες, αλλά είναι πολύ διαφορετικές, με διαφορετικά ονόματα και με διαφορετική επικεφαλίδα ε, και έτσι μεγάλη σύγχυση για τους πολίτες ε, οι οποίοι σε τελική ανάλυση απλά επιθυμούν μία λύση και δεν επιθυμούν να προσπαθούν πάση θυσία να ψάχνουν να βρουν πού να ξεκινήσουν ε, και πού να τελειώσουν. Έτσι λοιπόν, ενώ η Επιτροπή έλαβε βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση με ε, πρωτοβουλίες όπως είναι το ε, Your Europe, η πύλη αυτή που είναι πάρα πολύ καλό, αλλά και με μονομένα σημεία επαφής, εγώ πιστεύω παρόλα αυτά ότι υπολείπονται ακόμα πολλά. Κατόπιν τούτου στην έκθεσή μου προτείνω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να προσφέρει ένα και μόνο ζωντανό σημείο επαφής όπου κάθε κράτος ε, μέλος ε, μέσω του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μπορεί να δώσει συνέχεια στην όλη υπόθεση. Αυτές τις απόψεις συμπεριλαμβάνω στη ε, γνωμοδότησή μου. Βεβαίως, με μεγάλη μου χαρά ε, θα δεχόμουν την αντίδραση των συναδέλφων και προφανώς και τα σχόλιά τους. Αν επιθυμούν να καταθέσουν τροπολογίες ε, στη γνωμοδότηση αυτή, είναι σαφές ότι θα τις λάβω υπόψη μου. Και κάτι άλλο που αφορά στις, ε, προθεσμίες για την κατάθεση τροπολογιών είναι η 27η Μαρτίου και η ε, γνωμοδότηση πρόκειται να εγκριθεί από την Επιτροπή ε, στις 24 Μαρτίου. Σας ευχαριστούμε κύριε Μπουσουτήλ για την ε, παρέμβαση αυτή. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Κολίνσκι. Thank you very much, Madam Chair. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για τις προτάσεις που έχετε κάνει επί του ψηφίσματος της, για την έκθεση ΙΜΚΟ. Ο κ. Μπουσούτιλ έθνηση των δάκτυλων επί των τύπων των ύλων, εξήγησε τα προβλήματα και η Κομισιόν γνωρίζει τα προβλήματα αυτά και τώρα βέβαια με την όθηση αυτή θα διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας Πρόκειται για μία από τις πρωτοβουλίες που κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε την ανάγκη να διαφοροποιηθούν και να απλοπλασιαστούν οι πηγές πληροφοριών. Έχουμε λοιπόν μια πύλη εισόδου στο ίντερνετ για τις επιχειρήσεις και αυτή προσφέρει και την βοήθεια στις επιχειρήσεις, δηλαδή με εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης. Δίνει λοιπόν τη δυνατότητα αυτόματης εισόδου αυτή η πύλη. Είναι όμως ένα μόνο από τα πολλά εργαλεία που έχετε αναφέρει και για τις μελλοντικέ εκθέσεις η αναφορές που θα απευθύνονται στο Κοινοβούλιο, νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί η πύλη αυτή καθώς και άλλα μέσα. Υπενθυμίζω ότι το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Κομισιόν να εκδώσει την έκθεση αυτή για το Single Market Forum το περσινό. Αυτό θα επαναληφθεί φέτος, θα είναι η εβδομάδα, η δηλαδή της αγοράς Φέτος, το φθινόπωρο, κάθε πρωτεύουσα θα προωθήσει τρόπους για να προσεγγίσει η ενιαία αγορά τους πολίτες και να αποτυπωθεί ο τρόπος με τον οποίο βλέπουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις την ενιαία αγορά. Να διαπιστωθούν, να διαπιστωθεί μάλλον πού βρίσκονται τα κενά της ενημέρωσης και σε αυτά, βασισμένοι σε αυτά τα στοιχεία, θα προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπους για να κλείσουμε τα κενά αυτά. Οι προτάσεις που γίνονται σήμερα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών είναι πολύ θετικές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευχαριστώ θα τις λάβει υπόψη και θα τις επεξεργαστεί και επαναλαμβάνω ότι χαίρεται πολύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έκθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ τον εκπρόσωπο της Κομισιόν για την παρέμβασή του. Ο κύριος Γιάρη έχει το λόγο. Ευχαριστώ Σάιμον για τη σύνταξη εκθέσεως και φαίνεται πως το πέτυχες. Σπάνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έρχεται στην Επιτροπή Αναφορών και λέει ότι θα διπλασιάσει τις προσπάθειές της. Πολύ ωραία. Φαίνεται λοιπόν ότι όλοι κινούμεθα προς την ίδια κατεύθυνση. Και προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο. Βέβαια, καλό είναι να υπάρχουν δικαιώματα των πολιτών, αλλά πρέπει να είναι γνωστά και πρέπει επίσης να είναι και γνωστό πώς θα απαιτήσει κανείς την υλοποίησή τους. Συμφωνώ καταρχήν με το περιεχόμενο της έκθεσή σου, αγαπητέ Σάιμον, καθώς επίσης και με την υπόδειξη να δημιουργηθεί μια πύλη διαδικτύου που και οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να μπορούν ε, να αναζητούν τα δικαιώματά τους, αλλά επίσης να μπορούν να υποβάλουν και αναφορές. Γιατί εδώ στην Επιτροπή Αναφορών είμαστε λίγο ένας σεισμογράφος της διάθεσης των πολιτών. Δηλαδή θέλουμε αυτό το feedback. Αφενός λέμε ότι εντάξει έχουμε ταυτοποιήσει τα πράγματα, έχουμε νομοθεσίες, έχουμε κτλ. Αλλά θέλουμε και αυτό το λεγόμενο feedback, θέλουμε την αντίδραση των πολιτών δηλαδή, να δούμε πού υπάρχουν τα κενά, πού κάτι δεν λειτουργεί καλά, με τον κοινό στόχο πολίτες μας να αντιληφθούν την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα, ένα όλο όπου να αισθανόνται καλά να μπορούν να ζήσουν και να εργάζονται. Να υπάρχει επομένω μια αίσθηση δικαίου ασφαλείας ή μάλλον ασφαλεία δικαίου και αυτά είναι τα πράγματα που σε απασχολούν. Σε συγχαίρω λοιπόν και πάλι γιατί όπως είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να πολλαπλασιάσει τι προσπάθειές τη. άρα δηλαδή η επιτυχία τη εκθεσή σου είναι δεδομένη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γιάρ. Αν δεν ζητούν άλλοι συνάδελφοι τον λόγο, θα σας υπενθυμίσω απλώς ότι η κατάθεση τροπολογιών μπορεί να γίνει μέχρι τις 27 Τρίτου και διακόπτω την συνεδρίαση για 10 λεπτά.

Colleagues, I think that the 10 minutes are elapsed, so we can start. Ας αρχίσουμε γιατί πέρασαν τα 10 λεπτά του διαλύματος. Αναλαμβάνω τα ενία της ε, διευθύνσεως της συζητήσεως στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων για τα αποτελέσματα της ε, επίσκεψης στην Ρουμανία. Έχετε λάβει ένα πρώτο έγγραφο εργασίας που έχει συνταχθεί με την συνδρομή των υπηρεσιών. Να σας εξηγήσω τα διάφορα στάδια της αποστολής αυτής η οποία διεξήχθη στη Ρουμανία και διήρκεσε τρεις ημέρες. Προσπάθησα να μην ε, προβώ ιδιαίτερα σχόλια, να είμαι αντικειμενική. Και τα μέλη της ε, αντιπροσωπείας, τα οποία συνάντησαν την προηγούμενη εβδομάδα, συμφώνησαν. Γι' αυτό και το έγγραφο αυτό νομίζω ότι αντικατοπτρίζει πιστά τα σημεία από τα οποία όλοι συμφωνήσαμε. Έγιναν βέβαια παρατηρήσεις για τα διάφορα τμήματα του κειμένου και θα προσπαθήσω να απαντήσω συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τον κύριο Μποστινάρου. Ο κύριος Μποστινάρου μου έκανε κάποια αιτήματα για προσθήκη. Θα εξετάσω τα αιτήματα αυτά και θα προσπαθήσω να τα συμπεριλάβω στο κείμενο. Έλαβα επίσης ε, προτάσεις προσθήκης από τον συνάδελφο Πρέντα. που προστίθενται στα αιτήματα του κυρίου Χέφνερ. Στην ε, συνεδρία της προηγούμενης εβδομάδας που συζητήσαμε όλα αυτά τα θέματα, σε αυτή τη συνεδρία την οποία σας προανέφερα, έλαβα και κάποιες προτάσεις από τους συναδέλφους Έλμερ, Χέλμερ και Σαλαβράκο. Έχετε λοιπόν αναχείρας ε, το πρώτο σχέδιο. Ελπίζω να μπορέσω να το εμπλουτίσω και με τις δικές σας παρεμβάσεις σήμερα, ώστε η αποστολή αυτή, η επίσκεψη αυτή, να βοηθήσει και τις εργασίες μας που δεν, είναι, που δεν έχουν ως άλλο σκοπό από το να δίνουμε απαντήσεις στους συμπολίτες μας, να βρίσκουμε λύσεις αν βέβαια αυτό είναι δυνατόν, στα προβλήματα που τους απασχολούν, να είμαστε ενδιάμεση μεταξύ πολιτών και ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, όταν βέβαια αυτά ενέχονται άμεσα, ή είναι αρμόδια, καθήλυνα αρμόδια για τα ζητήματα των οποίων ε, επιλαμβανόμαστε εδώ στην Επιτροπή Αναφορών. Είχαμε διάφορες αναφορές, διαφορετικά θέματα και θα δείτε τις σχετικές λεπτομέρειες ε, στο σχέδιο έκθεσης. Προσπαθούμε να λάβουμε υπόψη όλες τις ε, διαπιστώσεις, ε, όλα τα συμπεράσματα στα οποία κατάληξαμε επιτόπου και να τα μεταφέρουμε στο κείμενο. Ουσιαστικά προσπαθούμε τώρα να οριστικοποιήσουμε το κείμενο και ελπίζουμε να βρεθεί μια λύση για τις αναφορές αυτές. Ελπίζω και να προσπαθήσουμε να μπορέσουμε να ε, διευκρινίσουμε και στους ε, συμπολίτες μας ε, όλα αυτά τα θέματα. Για τα πτηνά, για την οδηγία για τα πτηνά είχαμε ένα αίτημα από την πλευρά του αναφέροντος να μπορέσει να έρθει εδώ να παρέμβει. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο και στον εισηγητή και μετά, αν δεν έχετε αντίρρηση, μετά θα ξεκινήσει η συζήτηση. Θα έλεγα λοιπόν να δώσω ε, πρώτα απ' όλα τον ε, λόγο στην κυρία Μαρίνα Καζάκου, παρακαλώ. române reprezint una dintre Είμαι εκπρόσωπος της ε, ορνηθολογικής οργανώσεως και συγκαταλεγόμαστε μεταξύ ενός αριθμού μη κρατικών οργανώσεων που έχουμε ζητήσει να μην εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες ε, στην ε, περιοχή αυτή που εντάσσεται σε περιοχή Natura 2000. Πρόκειται για ένα αιωλικό πάρκο το οποίο αναπτύσσεται ε, ταχύτατα στην περιοχή αυτή της χώρας μας χωρίς καμία ξεκάθαρη στρατηγική. Τον Μάιο του 2011 υπήρχαν ήδη 4.000 ανεμογεννήτριες που επρόκειτο να εγκατασταθούν από τις οποίες 400 ήδη είχαν εγκατασταθεί τον Φεβρουάριο 2012 ο αριθμός των ανεμογεννητριών ανήρχεται σε 5.000. Ήδη από, δηλαδή προβλεπόμενες, ήδη 500 από αυτές είχαν ε, κατασκευαστεί και εγκατασταθεί. Από τις 500, συγγνώμη, από τις 5.000 που προβλέπονται συνολικά, 2.225 έχουν λάβει περιβαλλοντική έγκριση και θα κατασκευαστούν. Πολλές από τις ανεμογεννήτριες αυτές εγκαθίσταται ή πρόκειται να εγκατασταθούν σε περιοχή Natura 2000. Οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι κακοφτιαγμένες από επιστημονική άποψη. Δεν λαμβάνουν υπόψη ότι η περιοχή αυτή είναι περιοχή διόδου μεταναστευτικών πουλιών. Δεκάδες χιλιάδες πουλιά περνούν από την περιοχή αυτή στη διάρκεια της αποδημίας τους. Η ρωμανική Ντουβρουτζά, που είναι γειτονική με το βουλγαρικό έδαφος, είναι η μόνη περιοχή της Ευρώπης όπου απαντά τον χειμώνα ένα συγκεκριμένο είδος πουλιού σε αυτή την περιοχή υπάρχουν ήδη ή πρόκειται ακόμη να εγκατασταθούν πάνω από 500 ανεμογεννήτριες. Εκφράζουμε το αίτημα προς την Επιτροπή Αναφορών να πιέσει δηλαδή τις ρουμανικές αρχές ώστε να εκπονήσουν στρατηγική αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων επιπτώσεων δηλαδή στις περιοχές Natura 2000 των επιπτώσεων που θα προκύψουν από, αυτό, από την κατάσταση αυτού του αιωλικού πάρκου. Οι εργασίες θα πρέπει να διακοπούν μέχρι ότου αναπτυχθεί η στρατηγική αυτή και μέχρι ότου οριστεί σε ποιες περιοχές μπορεί να, μπορεί να εγκατασταθεί το αιωλικό πάρκο. Πριν ολοκληρώσω, θα ήθελα να πω ότι ορνηθολογική οργάνωση Ρουμανίας αλλά και οι άλλες οργανώσεις που συνυπογράφουν την αναφορά δεν είμαστε αντίθετοι με την μορφή της ολικής ενέργειας, αλλά θεωρούμε ότι δεν πρέπει να πέσει θύμα της προσπάθειας αυτής, των έργων αυτών, η περιοχή αυτή του Natura 2000, καθώς και το περιβάλλον γενικότερα. Πολύ ωραία. Στο σημείο αυτό ξεκινάει η συζήτηση, κυρία Χούκεν. Κοιτάξτε, πρέπει να σας πω ότι δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένη με αυτή τη διαδικασία δεν πήραμε την έκθεση και βλέπω ότι υπάρχει από τα τέλη Φεβρουαρίου. Και τώρα, αν κατάλαβα καλά, ήρθε την Τετάρτη στο Στρασβούργο, τότε που είχαμε πάρα πολλή δουλειά. Όπου έρχονται, έχουμε πλημμυρίδα ε, εγγράφων. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπόρεσα να το διαβάσω. Και θέλω να πω ότι αν είναι ε, πραγματικά αυτή η κατάσταση στη Ρουμανία και η Ρουμανία είναι σαν παράδεισο σε σχέση με την Βουλγαρία, εγώ δεν ξέρω, δεν πείθομαι. Έριξα μια επιπόλυτη ματιά, αλλά νομίζω ότι πραγματικά πρέπει να αναβάλουμε την εξέταση αυτής της υπόθεσης, γιατί απλά υπάρχει μια απάντηση από τις αρχές, υποτίθεται από απάντησε και η βιομηχανία, όλοι πάτησαν κανένα πρόβλημα αν αντιμετωπίζαμε με αυτό τον τρόπο την κατάσταση στην Βουλγαρία, η έκθεση στην οποία θα καταλήγουμε θα ήταν τελείω διαφορετική. Γιατί εκεί το ψάξαμε, προσπαθήσαμε να δούμε τι ακριβώ συμβαίνει. Θεωρώ λοιπόν ότι. Από ό,τι γνωρίζω, δεν είμαι ικανοποιημένη, κυρία Πρόεδρε. Δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένη με αυτό και νομίζω ότι ε, δεν μας προσέχετε. Ε, δεν ε, προσέχετε και δεν φροντίζετε την Επιτροπή. Λείπετε, δεν παίρνετε εκθέσεις, δεν δίνετε προτεραιότητα στα θέματά μας. Φοβάμαι δεν δίνετε προτεραιότητα στην Επιτροπή μας. Και είναι δύσκολο να κάνει κανείς τη δουλειά του αν δεν ε, στηρίζει ο πρόεδρος την Επιτροπή. Αυτό εδώ το έγγραφο ήρθε τόσο καθυστερημένα εσείς απλά είστε ο σύνδεσμος ανάμεσα στη βιομηχανία ε, και την Επιτροπή. Αυτό όμως δεν αρκεί. Και δεν είναι αυτός σωστός τρόπος ε, για να εργάζεται κανείς. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ να αναβληθεί αυτή η αναφορά. Είναι πολύ κακό που δεν ήρθαν οι άλλοι, οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, Πάντως ε, πρέπει να είμαι ειλικρινής, δεν είχα την ευκαιρία να ε, διαβάσω σε βάθος αυτή την έκθεση, όμως πρέπει να εκφράσω τη δυσαρέσκειά μου. Ο κύριος Ποστενάρο. Καταρχήν, κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι το σχέδιο έκθεσης αυτό έχουμε σήμερα μπροστά μας. Καλείται να απαντήσει μια σημαντική ερώτηση. Γιατί θα πρέπει η Επιτροπή Ναφορών να πάει και πάλι στη Ρουμανία. Και η μόνη απάντηση είναι ότι μέχρι σήμερα και από την τελευταία επίσκεψή μας βλέπουμε ότι δεν εφαρμόζεται στη χώρα αυτή οι νόμοι και οι διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε τόσες πολλές αναφορές ε, και κυρίως για ευαίσθητα θέματα όπως είναι το περιβάλλον, τα θεμελιώδη δικαιώματα, η ελευθεροτυπία και άλλα. Δεύτερον, υπάρχει ένα σημαντικό στοιχείο για πέντε ε, ευρωβουλευτές, εξαιρουμένων των Ρουμάνων ευρωβουλευτών δεν υπάρχει καμία σοβαρή αναφορά στα βασικά θέματα, στις ανησυχίες που εκφράστηκαν. Δηλαδή, γεωλογικός κίνδυνος, καμία απάντηση. Ευθύνη για το περιβάλλον, καμία απάντηση. Διάλογος ανάμεσα σε επενδυτές και κρατικές αρχές με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Ούτε και εκεί η απάντηση. Γιατί υπάρχουν τόσες πολλές ε, αντιρρήσεις ε, και στεναρή αντίδραση από την κοινωνία των πολιτών στη Ρουμανία, συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημίων, των ακαδημαϊκών κύκλων και γι' αυτό ε, δεν υπάρχει καμία απάντηση. Και τέλος, γιατί δεν αναφέρεται κάτι που αναφέρθηκε εδώ στην Επιτροπή των Αναφορών. Ε, μιλάμε για ένα χρυσορυχείο και χρειαζόμαστε ε, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτό το χρειαζόμαστε στην Επιτροπή μας για να είμαστε σίγουροι ότι η αξιολόγησή μας θα είναι σωστή και θα μπορέσουμε να ελέγξουμε την κυβέρνηση της Ρουμανίας κατά πόσον πράγματι εφαρμόζει την κοινοτική νομοθεσία ή όχι. Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Και ολοκληρώνοντας, θέλω να πω το εξής. Η καλύτερη απάντηση που μπορεί να δοθεί στις ανησυχίες μας ήταν πριν από μία εβδομάδα σε μία συνέντευξη του Υπουργού Περιβάλλοντος της Ρουμανίας όχι από την αντιπολίτευση, ούτε από την κοινωνία των πολιτών, ούτε από την Ακαδημία της Ρουμανίας. Ο ίδιος ο Υπουργός Περιβάλλοντος της, κυρίας, της Ρουμανίας, ο κύριος Μπόρμπεϊ, είπε σε μία συνέντευξή του, ναι πράγματι υπάρχει αυτή η διαδικασία ελέγχου του προγράμματος, όμως ε, δεν έχουμε ακόμα απάντηση και θέματα όπως ε, η βέλτιστη δυνατή υπάρχουσα τεχνολογία είπε επισκέφθηκα τη Σουηδία και τη Φινλανδία και είμαι τώρα πεπισμένος ότι το κλειστό σύστημα είναι το ασφαλέστερο και η Ρουμανία ε, θα αποτελέσει πρότυπο με έμπνευση από την ε, Σουηδία. Εμπνεόμενη από τη Σουηδία. Χρειάζεται μια απάντηση, αλλά η απάντηση δεν έχει ακόμα δοθεί. Κατόπιν, όσον αφορά την αποκατάσταση αυτού του χώρου, λέει ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει πολιτική συμφωνία τουλάχιστον και παραθέτω με ακρίβεια. Ε, να υπάρχει μέρημνα στον κυβερνητικό συνασπισμό. Πάνω από 100 τόσες χιλιάδες υπογραφές ε, ε, στάλησαν ε, με μία αναφορά στο Κοινοβούλιο της Ρουμανίας για το ίδιο θέμα και δεν είπε τίποτα από αυτού. Εγώ λοιπόν παραθέτω από την έκθεση και ευχαριστώ και πάλι την ειλικρίνεια της γραμματείας, για την, τη γραμματεία για την ειλικρίνειά της. Όταν ρωτήθηκε για τη στάση του, παραθέτω σελίδα 16, δεύτερη παράγραφος, που λέει ο ε, Γενικός Γραμματέας, ε, ο Υφυπουργός μάλλον, δέχεται ότι είναι υπέρ του προγράμματος αυτού, τέλος της παράθεσης. Τι άλλου είδους ε, παράδειγμα χρειαζόμαστε για μεροληπτική στάση αν ο αρμόδιος υπουργός δεν απαντάει στα θέματα και ο υφυπουργό που είναι αρμόδιος για την αξιολόγηση του προγράμματος ομολογεί ότι είναι υπέρ του προγράμματος. Πώς να αξιολογήσουμε και εμείς την αντικειμενικότητα σε αυτό το θέμα. Νομίζω ότι όλα αυτά ε, είναι σημαντικά και πρέπει να συμπεριληφθούν στην έκθεση για να διασφαλίσουμε ότι θα εισακουστεί η άποψη και η φωνή του αναφέροντος. Αυτή είναι η δουλειά μας, να εισακούεται η άποψη του αναφέροντος και όχι μόνο η άποψη του επενδυτή ή της κυβέρνησης. Και τέλος, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε εκπρόσωπος ε, του αναφέροντος ε, και της ορνηθολογικής εταιρείας. Η το θέμα είναι η κυβέρνηση της Ρουμανίας εφάρμοσε την κοινοτική νομοθεσία. Γιατί μας είπαν ότι δεν γνώριζαν ε, περί των ερευνών που έκανε η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Δεν είχαν ε, κανένα στοιχείο που να δείχνει ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία επί παραβάση. Αν λοιπόν δεν τα γνωρίζουν όλα αυτά, μπορούμε με κλειστά τα μάτια να δεχόμαστε την σοβαρότητα της αξιολόγησης. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να ακούσουμε και την άποψη της μιας πλευράς των αφέροντος και την άποψη της άλλης πλευράς των επίσημων εκπροσώπων, για να υπάρχει ισορροπία. Ε, θα καταθέσω μια σειρά τροπολογιών, όπως το έχω ήδη πει, και τελικά πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει και μια σύντομη πρόταση που να αφορά ε, στην ελευθερία των μέσων ενημέρωση. Γιατί αυτή η συνάντηση έλαβε χώρα, παρίσταντο πέντε ευρωβουλευτέ. Στο χώρο αυτό ήταν αρκετοί δημοσιογράφοι και αναφέροντες. Ε, όλοι αξιολόγησαν την κατάσταση των μέσων ενημέρωση και να μην αναφέρεται τίποτα από αυτό το βρίσκω λίγο περίεργο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι ε, θα μπορούσαμε να επιτύχουμε μια σοβαρή συνεργασία ανάμεσα σε όλες τις ε, πολιτικές ομάδες. Η κυρία Γκόντς, ε, ευχαριστώ. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να πάω μαζί στην αποστολή. Θυμούμαι όμως από προηγούμενες συζητήσεις τα θέματα που έχουν προκύψει από τις αναφορές. Γνωρίζουμε ότι ήταν περισσότερες από μία οι αναφορές αυτές. Εξετάζοντας το κείμενο, δεν βλέπω να προκύπτουν απαντήσει στις ερωτήσεις αυτές. Δεν είναι μόνο ρουμανικό το θέμα, γνωρίζοντα άλλωστε την ιστορία και το παρελθόν και τη περιβαλλοντική καταστροφή που έχει προκαλέσει λόγω και του χρυσορυχείου στη Ρώσα Μοντάνα, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο ξεπερνά τα ρουμανικά όρια. Μπορεί να επηρεάσει ολόκληρη την περιοχή και πολλές χώρες της περιοχής αυτής. Εγώ αναζήτησα απαντήσεις και εγγυήσεις ασφάλειας και δεν τις βρήκα. Είναι πολύ ε, αμφίδρομες οι γνώμες και από τις και οι γνώμες και τις κυβέρνησεις και των εμπειρογνωμόνων. Αλλά ο αρμόδιος ε, υφυπουργό για περιβαλλοντικά θέματα και σε μια χώρα όπου λαμβάνονται ελεύθερα οι αποφάσεις, νομίζω άνθρωποι στις θέσεις αυτές θα έπρεπε να μιλήσουν και για, την, για τη συγκρούση συμφερόντων. Γιατί κάποιο ο οποίο είναι αρμόδιο για το περιβάλλον πρέπει να, θέσει και, να καταθέσει και επιχειρήματα που υποστηρίζουν το περιβάλλον και όχι μόνο τις βιομηχανικές αυτές εγκαταστάσεις. Ίσως βέβαια εσείς γνωρίζετε περισσότερα γιατί εγώ μόνο τη γνωμοδότηση αυτή μπόρεσα να δω ίσως γνωρίζετε περισσότερο για το ποιες είναι οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά, αλλά δεν βλέπω ε, σοβαρές ενδείξεις ότι όντως γίνεται μια δημόσια διαβούλευση με συμμετοχή των ε, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, διότι πολλές οργανώσεις τέτοιες έχουν συλλέξει στοιχεία κλπ. Και ορισμένε από τις μελέτες, ε, μελέτες αναφέρονται στην έκθεση. Δεν τις γνωρίζω όμως εγώ. Δεν ξέρω εσείς αν τις γνωρίζετε και αν μπορεί κάποιος να τις αναγνώσει και να βγάλει κάποια συμπεράσματα. Αυτό βλέπω. Βλέπω περισσότερο να προβάλλονται επιχειρήματα, αλλά όχι επαρκώς θεμελιωμένα. Για, μιλάνε και για πυρηνικέ εγκαταστάσει. Κάτι το οποίο για εμένα μου προκαλεί έκπληξη, διότι διόλου δεν είμαστε πεπισμένοι ότι τα πυρηνικά εργοστάσια είναι πιο, τα πιο ασφαλή. Άλλωστε έχουμε και την, της, ε, την πρόσφατη εμπειρία της Φουκουσίμα. Νομίζω λοιπόν ότι πολλά θέματα παραμένουν ανοιχτά. Και νομίζω ότι όλα αυτά που διαβάζουμε εδώ δεν είναι πιστικά για να πούμε ότι όντω έχουμε τις απαντήσεις. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε την διαδικασία. Επίσης δε θα ήθελα να επανέλθω λίγο στο θέμα της ελευθερία των μέσων. Προφανώς, ή μάλλον φαίνεται να είναι, φαίνεται να είναι ξεχωριστό θέμα. Ωστόσο, συνδέονται τα θέματα αυτά, γνωρίζοντα ότι το κοινό λαμβάνει τι πληροφορίε του από τα μέσα είναι πολύ σημαντικό η ενημέρωση να είναι μη προκατηλημένη, να είναι απροκατάληπτη, να είναι δηλαδή ενήμερο το κοινό για να μπορέσει να λάβει τις αποφάσεις του για το αν θα θελήσει να παρέμβει, να διαμαρτυρηθεί κτλ. Δεν βλέπω όμως τα ρουμανικά μέσα να είναι και τόσο ελεύθερα, γνωρίζοντας τις δημοσίευσεις που έχουν γίνει για το έργο αυτό. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη και αυτό λοιπόν στην έκθεση, διότι εγώ όπως είπα δεν ήμουν παρούσα, γνωρίζω όμως ότι υπήρξαν συναντήσει με δημοσιογράφου. Δεν είναι εντελώς ξεχωριστό το θέμα, είναι πολύ στενά συνδεδεμένο. Οι πληροφορίε δηλαδή που μπορεί να έχει στη διαθεσή το κοινό για τέτοιου είδους έργα. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε ακόμα πολλή δουλειά να κάνουμε για την έκθεση αυτή και δεν θεωρώ, άλλωστε προέρχομαι από γειτονική χώρα και χώρα η οποία έχει πληγεί σοβαρά από την περιβαλλοντική καταστροφή για την οποία μιλούμε. Νομίζω δεν είναι επαρκής οι απαντήσεις. Θα ήθελα κύριε Πρόεδρε Äh, Κοιτάξτε, καταρχήν ε, το βρίσκω καλό το ότι αυτές οι επισκέψεις μας, οι επιτόπου επισκέψεις, ε, τελικά εξελίσσονται σε μια πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση. Ε, Βεβαίω, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, πρέπει να πω ότι όσον αφορά τη Ρουμανία, στο Βερολίνο δεν συμφώνησαν όλοι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι για την ύπαρξη ενός και μόνο εγγράφου. Όπως ε, αυτά που είπες για την κυρία Ματσόνη, ε, δεν ήταν σωστά, δεν σωστό αυτό που της είπε. Στη δημοκρατία, ε, όταν κατήθε μια πρόταση, αυτό αποτελεί τη βάση διαπραγμάτευσης. Κάπου πρέπει κανείς να ξεκινήσει. Το λέω απλώς αυτό, Σε αυτή λοιπόν τη διαδικασία δεν φταίει η επικεφαλής αντιπροσωπείας για αυτό το έγγραφο. Κάπου πρέπει να γίνει κάποια αρχή. Δεν ήταν σωστό αυτό που έκανες προηγουμένως. Αυτό θέλω να πω είναι το ένα. Το δεύτερο. Αυτή είναι η εντύπωσή μου γιατί κατά νου έχω την επίσκεψη στο Βερολίνο. Θα υπάρξει και για αυτήν έκθεση. Και το θέμα είναι πρέπει να συμφωνήσουμε ε, τι θα, κάνουμε και τι πρέπει να κάνουμε με τις επιτόπιες εκθέσεις. Γίνεται η έκθεση, υπάρχουν οι επίσημοι, οι ανεπίσημοι μετέχοντες ε, από τις χώρες όπου γίνεται η επίσκεψη και μετά κατατίθεται μία έκθεση και η έκθεση αυτή ψηφίζεται στην Επιτροπή. Και στην έκθεση μπορεί να, συμπεριλαμβάνεται μόνο, να συμπεριλαμβάνονται μόνο αυτά που έλαβαν χώρα. Η αντιπροσωπεία που επισκέφθηκε τη χώρα, έκανε μερικά πράγματα, αλλά δεν μπορούμε εμείς στην έκθεση να γράψουμε πράγματα που δεν έχουν λάβει η χώρα. Και παρόλα αυτά, όταν είμαστε εδώ και ψηφίζουμε για κάτι, ενδέχεται σε ορισμένα σημεία οι αποφάσει που λαμβάνονται να είναι πλειοψηφικέ. Ενδέχεται λοιπόν να υπάρχουν εκθέσεις ε, όπου κάποιοι βουλευτές να λένε και να μπορούν να πούν ότι εγώ δεν συμφωνώ με αυτό το θέμα. Αυτά νομίζω πρέπει να τα ξανασυζητήσουμε και στην, κυρίως στη συνάντηση των συντονιστών. Το πώς δηλαδή συντάσσονται οι εκθέσεις και πώς ολοκληρώνονται. Σας το λέω. Ε, με την έκθεση του Βερολίνου διαπιστώσαμε ότι η κατάσταση δεν είναι τόσο απλή. Γι' αυτό λοιπόν εγώ προτείνω στις συνεδρίες των συντονιστών να αποφασίσουμε πώς θα προχωράμε. Και τέλος, θεωρώ ότι η Επιτροπή είναι εκείνη που αποφασίζει. Αυτό όμως που κατατέθηκε είναι μία πρόταση. Και δεν πρέπει να κρεμάμε αυτούς που φέρνουν την είδηση, Απλώς μας ήρθε εδώ η είδηση και με τη Ρουμανία προχωρήσαμε πιο πολύ από ότι με το Βερολίνο. Δεν είμαστε και πολύ ευχαριστημένοι, αλλά είναι μια αρχή ε, και εγώ ε, ευχαριστώ την ε, Πρόεδρο που έκανε αυτή την αρχή. Υπάρχουν άλλοι που επιθυμούν να λάβουν το λόγο, παρακαλώ. Λοιπόν, κοιτάξτε, προφανώς θα συγκρουστούμε και πάλι για το έγγραφο αυτό. Αυτό απλά είναι σχέδιο γράφου, το έχω συζητήσει και με άλλους που συμμετείχαν στη, στη συνάντηση. Αυτό το έγγραφο απλά είναι ε, μια παρήθμιση των επισκέψεων. Ε, βεβαίως, ε, καλό είναι να ασκείται κριτική, αλλά αν ήταν πιο επικοδομητική η κριτική θα μου άρεσε καλύτερα. Πρέπει να σας πω και το λέω αυτό από τη συνάδελφο κυρία Γκόνς, ότι ε, δεν ε, θεωρώ ότι μέσα στην έκθεση αναφέρουμε ότι είμαστε ευχαριστημένοι ότι έχει ολοκληρωθεί η δουλειά. Κάτι άλλο. Υπάρχει ε, η ανάλυση των υπέρ και των κατά που εντοπίσαμε κατά τη διάρκεια των τριών ημερών της επισκεψής μας. προσπαθήσαμε λοιπόν να καταγράψουμε τις ε, ε, πληροφορίες που πήραμε και σας λέω ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να βελτιωθεί η έκθεση. Δεν είχα το χρόνο για να συμπεριλάβω τις ε, απόψεις του σαντέλφου Μποστινάρου. θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας πριν φτάσουμε στην, στην κατάθεση τροπολογιών. Γιατί αυτό θα γίνει, αλλά Καταρχήν είχαμε πει ότι θα συμφωνήσουμε επί της μεθόδου και νομίζω είχαμε συμφωνήσει ότι θα υπάρξει και άλλη μία συνάντηση για να ε, καταλήξουμε σε ένα έγγραφο περισσότερο αποδεικτό. Ε, τώρα, όσον αφορά το θέμα για τα μέσα ενημέρωσης, πρέπει να πω ότι αυτό είναι ένα θέμα που αφορά τους συντονιστές. Η έννοια του ε, ε, το θέμα του προγράμματος μιας επίσκεψης εγκρίνεται από τους συντονιστές. Εγώ ως πρόεδρος ε, απλά τηρώ ένα πρόγραμμα που δεν ε, προέβλεπε τη συνάντηση με τους ε, αναφέροντος ε, σχετικά με την οργάνωση πληροφοριών στη Ρουμανία. Ορισμένα μέλη της Επιτροπής, κυρίως ο κύριος Μποστινάρου, εξιοφύσιο είχε κάποια συνάντηση και νομίζω όποιος ευρωβουλευτής ήθελε μπορούσε να συναντήσει επιτόπου όποιον ήθελε και να τοποθετηθεί αλλά Θεωρώ ότι ο κύριος Μπεστινάρου και θα συμφωνήσει είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Μέσα στην έκθεση να ε, ένα θέμα το οποίο δεν προβλεπόταν στο πρόγραμμα και εγώ βεβαίως ε, δεν μπορώ να πω ότι είχα υπόψη μου ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Επαναλαμβάνω, εν πάση περιπτώσει, επειδή τα προγράμματα των επισκέψεων τα αποφασίζουν οι συντονιστές. Είναι δική τους κυρίαρχη θέληση να επαναφέρουν το θέμα αυτό, ακόμα και αν δεν προβλεπόταν στην ε, συνάντηση. Για μένα, τέτοιου είδους εργασία, ε, είμαι πολύ ευέλικτη απέναντι σε τέτοιου είδους ε, εργασία, ε, δεν νομίζω ότι πρέπει να τσακωνόμαστε μεταξύ μας, πρέπει να είμαστε κοντά στους πολίτες. Και εάν τελικά από τα ε, διάφορα στοιχεία που συγκεντρώνουμε καταλήγουμε στο ότι μπορούμε να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα, αν υπάρχει λοιπόν κάτι συγκεκριμένο, ε, θεωρώ ότι αυτό πράγματι πρέπει να το κάνουμε. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι όλοι έχουν το δικαίωμα, αλλά και την υποχρέωση να ε, ασκούν πολιτική. Αλλά όπως λέμε και πολύ συχνά, αυτή ακριβώς ε, είναι η επιτροπή όπου πρέπει να περιορίσουμε στο ελάχιστο την άσκηση πολιτικής. Δεν είναι αλήθεια αυτό που λέει η συνάδελφος κυρία Χόκεν, ότι απλά παρατηρώ ε, το τι γίνεται. Και η κυρία Χόκεν που κι άλλη φορά με έχει επικρίνει να πει κάτι συγκεκριμένο και εμείς και η Γραμματεία θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Κλείνει λοιπόν το σημείο αυτό και τελειώνουν οι εργασίες μας ε, και στις 5.30 ε, θα έχουμε τη συντάνηση των, ε, συνάντηση των συντονιστών. Κτό βέβαια αν θέλουν οι συνάδελφοι να ξεκινήσουμε τώρα τη συνάντηση των συντονιστών. Να ξεκινήσουμε νωρίτερα. Μετά από πέντε λεπτά. Γεια σας.